της Ευρώπης. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις ε, ψηφοφορίες. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, απαλλαγή για τον Γενικό Ευρωπλογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης του 2009, Επιτροπή. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, λέει η πρόεδρος. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία την απόφαση παριθμών 2. Είναι οργανισμός ε, για, ε, για τον πολιτισμό. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται υπαριθμών 3 εκτελεστική επιτροπή για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία έκλειση ψηφοφορία Εγκρίνεται απόφαση παριθμών 4 για την Εκτελεστική Επιτροπή για την Υγεία και τους Καταναλωτές. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εκτελεστικός οργανισμός ε, για τα συνοριακά, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ε, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται εκτελεστικός οργανισμός του, Συμβουλίου, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έρευνα ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εκτελεστικός οργανισμός για την έρευνα. Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Παράγραφος 78. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 79. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 80. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλω παρακαλώ να μου στείλετε ένα τεχνικό γιατί δεν μπόρεσα να ψηφίσω κατά. Παράγραφος 81 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 82. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα, τροπολογία υπαριθμών 5 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 6. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία περιθμών 4 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Για την 10. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος ως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα, στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται η ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Χατζημαρκάκη, ειδικέ εκθέσεις ε, του ε, Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2009 της Επιτροπής. Ψηφίζουμε για την 51, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 61 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Για το σύνολο της πρώτας ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία ε, ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σχεδόν ομόφωνα ψηφίστηκε η έκθεση αυτή. Τώρα, η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφορία για την έκθεση του κυρίου Ήταλα για την απαλλαγή για το 2009, Γενικός προεπιλογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εξετάζουμε λοιπόν την πρόταση λήψης απόφασης, ε, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ξετάζουμε τώρα την ε, πρόταση ψηφίσματος, ε, τροπολογία υπαριθμών 1, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μισό λεπτό. Εγκρίνεται, εγκρίνεται λέει η πρόεδρος τώρα. Ψηφίζουμε ε, την τροπολογία περιθμόντρια 3, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Καταπίπτει η τροπολογία περιθμών 2. Τροπολογία υπαριθμών 5 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, μοιάζει να έχει εγκριθεί. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την υπαριθμον... τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 86. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 87 σε έξι διαφορετικά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, πέμπτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, έκτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 90. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 16 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8, ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 9. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Votazione chiusa. Respinto. Απορρίφθηκε. Η 17. Η τροπολογία με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 18 η τροπολογία, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Τροπολογία 10, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 119. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129. Παράγραφος. Τροπολογία προφορική της κυρίας Λούλινγκ Κυρία Λούλινγκ, κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους ομάδας μου θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία για την παράγραφα αυτή. Πρόκειται για μια τεχνικής φύσεως μάλλον τροπολογία που δεν είναι όμως καθόλου ανώδυνη. Θα πρότεινα λοιπόν τα δύο και τρία γιώτα για, αυτές, για αυτά τα δύο εδάφια, δεν ξέρω γιατί τα λένε ΙΙ και ΙΙ, ο μέλλοντας να αντικατασταθεί από αόριστο. Δηλαδή, τα μέτρα που αναφέρονται στα δύο αυτά εδάφια εφαρμόστηκαν εδώ και καιρό. Ε, πάει μια διετία που ισχύουν. Δεν έχει λοιπόν νόημα να ζητούμε ορισμένα μέτρα για το μέλλον από τη στιγμή που τα μέτρα αυτά ήδη ισχύουν. Νομίζω ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε την κοινή λογική και να αντικαταστήσουμε το μέλλοντα από τον αόριστο. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν σημειώνει τη δυνατότητα ε, περιορισμένης σύνταξης από τα 50 χρόνια και δυνατότητα να, να, λάβει κανείς ένα κεφάλαιο που αναφέρονται σε 25 χρόνια ε, συντάξιμα, καταργήθηκαν. Γιατί η συντάξιμη ηλικία πέρασε από τα 60 στα 63 και οι διαχειριστές του Ταμείου προσκλήθηκαν να να εγκρίνουν κτλ. Όλα αυτά τα μέτρα ήδη έχουν ε, θεσπιστεί και ήδη ισχύουν. Δεν χρειάζεται μέλλοντας πια εδώ. Ωραία, ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, να ψηφίσουμε. ποιο είναι υπέρ. Μια στιγμή, μια στιγμή γιατί θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία κατά τη για το πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και τώρα το δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 130. Κατά τμήματα, σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν σηκώστε όλοι τα χέρια. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονική. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 131, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 132, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται τρίτο τμήμα προτιμάται ηλεκτρονικό έλεγχο καλώς άρχεται η ψηφοφορία τέλος απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα τρίτο τμήμα τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, καλώς, αλλά καλύτερα σηκώτε τα χέρια για να κερδίσουμε χρόνο. Άρχεται η ψηφοφορία για το τρίτο τμήμα. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 133. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 142 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα το σύνολο Τη έκθεση του ψηφίσματο όπω έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μα. Έκθεση Ριβελίνη για την απαλλαγή διαχειριστική χρήση 2009, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 4 της πρώτης ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρα, ε, τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Κατά τμήματα έχουμε 7 χωριστά τμήματα. Με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται έκτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και έβδομο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος, όπως έχει τροποποιηθεί, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Ριβελίνη. Απαλλαγή 2009, Γενική ε, Γενικός Προϋπολογισμός Ένωσης, ελεγκτικό συνέδριο, επόμενη έκθεση. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρόταση απόφασης. Τώρα περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. η ψηφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της πρώτας ψηφίσματος ως με ονομαστική κλίση. Ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ε, πρόκειται για τον κύριο Ριβελίνη. Απαλλαγή για το 2009. Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ψηφίζουμε τώρα ε, με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ε, ξετάζουμε λοιπόν την πρόταση ψηφίσματος. Και ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 3 σε ε, ξεχωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, ε, κατά, αποχές ε, μοιάζει να απορρίπτεται η πρόταση αυτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπερθμών 4, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Παρακαλώ να σηκώσετε τα χέρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ε, σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Από ό,τι βλέπω όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την 7. Ε, Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, μοιάζει να απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Η τροπολογία υπαριθμών 8. Ψήφι πρέ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η εννέα με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Respinto. Ε, Απορρίπτεται. Η 11 ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 1. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα παρακαλώ η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Πάντα έκθεση Ριβελίνη, απαλλαγή 2009, Γενικό προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή των Περιφερειών. Ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματο με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται εξετάζουμε την πρόταση ψηφίσματος. Η τροπολογία υπαριθμών 1 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 3 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο της πρώτας ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι κύριε Σιγητά. Έκθεση ΣΤΑΣ. Απαλλαγή για το 2009, 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Θέτω σε ψήφιστο σύνολο με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, εξετάζουμε την πρόταση ψηφίσματος και θα ψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 2. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μητροπολογίες 1 και 3 ταυτόσιμες ψήφι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Έκθεση Σταυρακάκη. Απαλλαγή 2009. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ισηγητά. Τώρα όμως θα πρέπει να εγκρίνουμε την πρόταση ψηφίσματός σας και θα ψηφίσουμε την τροπολογία παριθμών 1. Ψηφί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 3 υπέρ. Κατά αποχές Φαίνεται να έχει εγκριθεί, αν θέλετε να την ελέγξουμε όμως. Δεν θέλετε. Προχωρούμε. Η τέσσερα τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι μου φαίνεται ότι έχει απορριφθεί όμως τώρα. Σηκώνετε χέρια σας παρακαλώ. Ε, τώρα ελέγχουμε την τροπολογία υπερθμών 4 ηλεκτρονικά. Άρχισε η ψηφοφορία. Τελείωσε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμό 5. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμό 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 11 υπέρ κατά αποχές φαίνεται να έχει απορριφθεί. Θέλετε έλεγχο? Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 11. Πέρασε. Approvato, però io Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ψηφίζετε. Η 12 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 υπέ. κατά άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 10 ψήφι υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε με ανομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Σταυρακάκι. Όλο λάθος σας λέω. Ε, τώρα, Οργανισμός Εμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την απαλλαγή 2009. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. πέρας. Εγκρίνεται. Εξετάζουμε το σχέδιο ψηφίσματο. Χωρί τροπολογίε. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση τώρα. η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Κύριε Στραβρακάκη. Σταβρακάκη, εν πάση περιπτώσει. Για την απαλλαγή τώρα της κοινή επιχείρηση για τον ΙΤΕΡ και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύνδεξης. Pongo in votazione per appello nominale, Ανομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρασε. εγκρίνεται. Πρόταση ε, ψηφίσματος χωρίς τροπολογίες, ονομαστικά, αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Ε, προχωρούμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Μορέιρα για το Πακιστάν. Εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτη ανάγκης. Με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε την τροπολογία 43. Άρχεται τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 31... τροπολογία τροπολογίες Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Τις ψηφίζουμε μαζί. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία 12 με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Ο κύριος Μπιντεγκάν προτείνει μια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε. Στο 2 του 9α, ε, εκεί που λέμε ε, κατέτηση κράτους μέλους, θα θέλαμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που δρά εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Θέλουμε να γίνει συμβατός αυτός ο κανονισμός με άλλες ασφαλιστικές δικλείδε, όπως ε, η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Νότια Κορέα. Θέλουμε ευθυγράμμιση των διαφόρων κειμένων. Ευχαριστώ. Ci sono obiezioni αντιρρήσει. υπάρχουν αντιρρήσει από ό,τι βλέπω όχι, κατόπιν τούτου μπορούμε να προχωρήσουμε. Ψηφίζουμε για την ε, τροπολογία υπερθμών 33, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 42, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την ε, τροπολογία 34 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 38 υπέρ παρακαλώ. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Μάλιστα. Για την 34 ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38, παρακαλώ να σηκώσει τα χέρια, ψηφίζουμε παρακαλώ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 40, υπέρ. Η 39 πρέπει να ε, σηκώσετε τα χέρια. Ε, πρέπει λοιπόν να σηκώσετε τα χέρια. Μισό λεπτό. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Τροπολογία 40. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 41 ε, ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 44 σε ξεχωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ε, αποχές ε, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 45 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για την πρόταση της Επιτροπής ως τροποποιήθηκε υπέρ κατά εγκρίνεται ο κύριος Μορέιρα θέλει να παρέμβει Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου έχω εντολή από την Επιτροπή μου να ζητήσω την αναβολή της ψηφοφορίας επί του νομοθετικού ψηφίσματος Αυτό άσχετα με την ε, δική μου την προσωπική θέση για το θέμα αυτό, το ζητώ ως εκπρόσωπος, ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Μισό λεπτό, πρέπει να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. συμφωνούμε με την πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Επομένως μπορούμε να ψηφίσουμε για την πρόταση του κυρίου Μορέλα. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής κατά, άρα η πρόταση έγινε δεκτή και θα υπάρχει μια επιστροφή, επαναπομπή στην, ε, στην Επιτροπή. Έκθεση του κυρίου Σούτλερ για τις ε, με τα μεταβατικέ διατάξει που αφορούν τις διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις τρίτες χώρε και αφορούν τι επενδύσει. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Σηκώστε το χέρι σα, ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιο είναι κατά. αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Το αντίστοιχο σημείο. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε, θέλετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία η τροπολογία 4. Υπέρ. Ε, άρχεται η ψηφοφορία προφανώς. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1, το αντίστοιχο σημείο, ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1, το αντίστοιχο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Και κόντρο. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Πάλι το αντίστοιχο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μήπως ε, θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν σηκώνετε το χέρι σας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέραση Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Ε, δεν μπορώ να εκτιμήσω το αποτέλεσμα όσα έχει, άρα θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σηκώσετε το χέρι σας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1, το αντίστοιχο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, πάλι το αντίστοιχο τμήμα του εκτιμώντας 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, θέτουμε σε ψηφοφορία την πρόταση επιτροπής όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Θα το προσψηφίσει το, το, το κείμενο πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και συγχαίρουμε τον ε, εισηγητή. Λοιπόν, έκθεση του κύριου Μορέιρα για την μακροοικονομική ενίσχυση προς την Γεωργία. Τρεις τροπολογίες τις ψηφίζουμε από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Επομένως, θέτω σε ψηφοφορία το τροποποιημένο κείμενο της Επιτροπής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Αρχίζει η ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρα της ψηφορίας Εγκρίνεται. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. Περνάμε τώρα στις ε, δηλώσεις, ε, στις επεξηγήσεις ψήφου.